Η ψηφοφορία για την έκθεση Μάρτιν θα γίνει την Τετάρτη και η επόμενη Σύνοδος Ολομέλειας θα συνέλθει από το πρωί από τις 9 μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι ε, τα μεσάνυχτα. Έχετε την ημερήσια διάταξη στα έγγραφα της Συνόδου και στην ιστοσελίδα. Λύεται η συνεδρία.